Καλώ ήρθατε στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σημείο πρώτο, έγκριση της ημερήσια διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια από την πλευρά σα, τότε μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο σημείο 2. Συνάδελφοι, η συνεδρίαση αυτή έρχεται αμέσως μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι και η ακροτελεύτια συνεδρίαση τη Επιτροπή ΑΦΕΤ αυτή τη θητεία. Συγχαίρω όλου του ε, συναδέλφου που εξελέγησαν και χαίρομαι που θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα και στην επόμενη θητεία. Και επίση να ευχαριστήσω και όλου του συναδέλφου που θα επιστρέψουν για την αφοσίωσή του και τη σκληρή του δουλειά στα πλαίσια αυτή τη Επιτροπή. Και ελπίζω να έχουμε τη στήριξή του και στα μελλοντικά μα ε, βήματα. Έχουμε πολύ ε, λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 12.30. Οπότε να ξεκινήσουμε αμέσως και περνάω στο σημείο 3. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Γιωχάνης Χάν, ο οποίος κάθεται ακριβώς δίπλα μου. Είναι εδώ για να μας παρουσιάσει το, τις πρόσφατες εκθέσεις όπως εγκρίθηκαν για την διεύρυνση. Ε, θα μας παρουσιάσει τις αναχώρα εκθέσεις. Πρωτού δημοσιοποιηθούν και τις παρουσιάσει και στο κοινό. Πρώτα το Κοινοβούλιο και μετά δημοσίω. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να ενημερωθεί εγκαίρως ώστε να μπορέσουν και οι βουλευτές να ασκήσουν τα καθήκοντά τους την εξέταση και την έγκριση της όλης διαδικασίας της διεύρυνσης. Θα καλέσω τους συναδέλφους μου από το Ευρωκοινοβούλιο να και να τους ευχαριστήσω μάλλον ε, και να τους καλωσορίσω γιατί μετά την ε, πολύ φορτωμένη, το φορτωμένο πρόγραμμά τους μετά τις εκλογές ε, κατάφεραν να συμμετέχουν σε αυτή την έκταση συνεδρίαση. Έχουμε 7 χώρε να εξετάσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γι' αυτό θα σα παρακαλέσω να περιοριστείτε στα 15 λεπτά, κύριε Χάν, ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο και για, την, για το διάλογό μα μετά. Θα ήθελα να θυμίσω επίση στου συναδέλφου ευρωβουλευτέ ότι η σημερινή συνεδρίαση αφορά την παρουσίαση απλώ των εκθέσεων. Θα ακολουθήσουν πολλέ ανταλλαγέ απόψεων για το θέμα τη κάθε χώρα ξεχωριστά του ερχόμενου μήνε βάσει τη τακτική διαδικασία. Οπότε θα είμαι πολύ αυστηρό στο χρόνο αγόρευση σήμερα. Καταρχά, να δώσω το λόγο στους, θα δώσω το λόγο στου συντονιστέ και του ε, αρμόδιου και του προέδρου αντιπροσωπιών. Ε, Σα ε, δίνω το λόγο, κύριε Χάν. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, εισαγωγή σου που ήταν σημαντική. ορίζω τους παλιούς φίλους και χαίρομαι που υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές. Λοιπόν, να περάσω στο θέμα. Πριν από 3,5 μόλις χρόνια, τον Νοέμβριο του 2015, ήρθα στο σώμα σας για να σας παρουσιάσω την μέσο πρόθεσμη στρατηγική την, ε, της ε, πολιτικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα τη στρατηγική της Επιτροπής πρόσφατα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας για να υπάρξει μια σταθερή και δίκαιη πολιτική διεύρυνση στην τελευταία πενταετία και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι και πάλι εδώ για να παρουσιάσω το πακέτο διεύρυνσης ε, για αυτή την χρονιά Από ό,τι έμαθα, καθοδόν ενεκρίθη επισήμως και από την Επιτροπή, οπότε το πακέτο που σας παρουσιάζω είναι επίσημο. Το φετινό πακέτο κάνει απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί, παρουσιάζει την κατάσταση πραγμάτων και την ε, πρόοδο που έχουν επιτύχει οι υποψήφοι για να πληρώσουν τα κριτήρια. Μπορούμε να πούμε ότι στα Δυτικά Βαλκάνια έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα λόγω τη συγκεκριμένη προσπάθεια μα. Είχαμε την πρώτη συνάντηση κορυφής με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων για 15 χρόνια. Σωστά σημειώνει και χαιρετίζει την πρόοδο. Ορισμένη, σε ορισμένες περιπτώσει ε, καταπληκτική πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Αλλά υπάρχουν ακόμη προκλήσεις και το πακέτο τονίζει και τι ανεπάρκειες και δίνει και οδηγίες. Αυτό αποδεικνύει την αξιοπιστία της Ένωσής μας και την δυνατότητα που έχει να επηρεάζει την κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε και εμείς να επιτύχουμε την πρόοδο που αντιστοιχεί ε, στην πρόοδο που επέτυχαν οι εταίροι μας και για την Αλβανία και για την Βόρεια Μακεδονία η Επιτροπή επαναλαμβάνει την ε, πρότασή τη, τη σύστασή τη, ε, την περσινή προ το Συμβούλιο να ξεκινήσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Υπάρχουν προβλήματα όμω στην περιοχή. Οι υποψήφιε χώρε κατά προτεραιότητα πρέπει να έχουν πιο βιώσιμα αποτελέσματα σε διάφορα θέματα κλειδί. Πρώτα απ' όλα το κράτο δικαίου. Από κάθε άποψη. Δεύτερον, ο κύριο στόχο τη πολιτική μα διεύρυνση είναι να συνεχιστεί η εξαγωγή τη σταθερότητα. Δεν θα εισαγάγουμε τι διμερεί διαμάχε και την αστάθεια που αυτό θα ε, είχε ως συνέπεια. Γι' αυτό τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να επιτύχουν περισσότερη πρόοδο για τη συμφιλίωση, καλές σχέσεις γειτονίας και περιφερειακή συνεργασία εμπνευσμένη από το παράδειγμα της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας. Τρίτη σημαντική πρόκληση, η οικονομία. Η οικονομία των χωρών αυτών έχει ακόμη σημαντικές δομικές αδυναμίες. Για να αξιοποιήσουν τι δυνατότητε Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερε μεταρρυθμίσει, να μειωθεί η ανεργία. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπιστούν και οι δημογραφικέ προκλήσει, γιατί είναι χαμηλή γεννητικότητα και μεγάλη μετανάστευση. Πρέπει λοιπόν να ανέβει το βιωτικό επίπεδο των λαών. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται περιφερειακή ενοποίηση. Η πρόσφατη συμφωνία για την περιαγωγή στην περιοχή που υπεγράφει από τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι παράδειγμα καλής περιφερειακής συνεργασίας που θα έχει ουσιώδη ωφέλη και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Να υπογραμμίσω το εξή σημαντικό. Η Ένωση, κατά πολύ, είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρο των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την δραστηριότητα στον επιχειρηματικό και μεδετικό τομέα τη Κίνα που αυξάνεται. Αυτό δίνει ευκαιρίε. αλλά οι επενδύσει αυτέ πολύ συχνά αμελούν το κοινωνικό, το κοινωνικο κοινωνικο-οικονομικό ε, θέμα και την βιωσιμότητα της οικονομίας των περιοχών. Γι' αυτό πρέπει να αυξηθεί η αντοχή της περιοχής σε οποιασδήποτε αλλαγές και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή πρέπει να σέβεται τις προδιαγραφές της Ένωσης. Ποια είναι τα κύρια ευρήματα για τις χώρες επιμέρους. Οι χώρες ανταποκρίθηκαν στις ευκαιρίες που τους δίνει η στρατηγική μας για τα Δυτικά Βαλκάνια με καλό τρόπο. Ιδιαίτερα με χαροποιεί η προσπάθεια που γίνεται στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Στην Αλβανία γίνεται μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, μια αξιολόγηση των δικαστών και εισαγγελέων. Η Βόρεια Μακεδονία συνεχίζει το φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, αλλά έχει και αυτή την ιστορική συμφωνία με την Ελλάδα που έλυσε το πρόβλημα τη συμφωνία που είχαμε για τόσο καιρό. Και η διμερή τη συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι υπόδειγμα επίση πώ μπορεί να αυξηθούν οι καλέ σχέσει γειτονία σε όλη την περιοχή. Είναι λαμπρό παράδειγμα για τι ε, χώρε συνολικά τη περιοχή και είναι σαφή ένδειξη τη ε, ισχύω τη Ένωση και του παραδείγματό τη. Και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018 ομόφωνα ε, κατέληξε σε πορίσματα και η Επιτροπή προτείνει τώρα να ξεκινήσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει και με την Αλβανία και με τη Βόρεια Μακεδονία. Για να παραμείνουμε αξιόπιστοι, πρέπει να σεβαστούμε τι δεσμεύσει μα, να ανταποκριθούμε θετικά όταν οι χώρε επιτυγχάνουν τι δικέ του δεσμεύσει. Υπάρχει πρόοδο ε, σε διάφορα θέματα, αλλά το Μαυροβούνιο και η Σερβία πρέπει να κάνουν περισσότερε προσπάθειε σε ζωτικού τομεί. Χρειάζονται να εφαρμόσουν επιγόντω μεταρρυθμίσει για το κράτο δικαίου αυτός είναι ο πιο σημαντικός τομέας και η πιο σημαντική προϋπόθεση για να προχωρήσουν στην ευρωπαϊκή οδό τους. Πρέπει να επιτύχουν οπωσδήποτε την πρόοδο που χρειάζεται στα κεφάλαια 23 και 24 για το κράτος δικαίου. Ο διάλογος Βελιγραδίου και Πρεστίνας πρέπει να δημιουργήσει ένα κατάλληλο κλίμα για την ολοκλήρωση μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ανταμείψει συγγνώμη, όχι, να τιμωρήσει οποιασδήποτε προκλητικές ενέργειες. Το κοσυφοπαίδιο πρέπει να επανέλθει στην πρόοδο προ την Ευρώπη. Το Βελιγράδι έχει επιτύχει κάποιε προσπάθειες, αλλά συγγνώμη, η Πριστίνα έκανε μερικές θετικέ προσπάθειες, αλλά οι δασμοί που επέβαλε στα προϊόντα από τη Σερβία και την Βοσνία-Ζεγοβίνη ήταν πολύ αρνητικό βήμα. Η Επιτροπή επίση σήμερα ενέχρινε την γνωμοδότησή της για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και για την αίτησή της ε, να ενταχθεί στην Ένωση. Η γνωμοδότησή μας δίνει συνολική κατεύθυνση για να βελτιωθεί η κατάσταση στο κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ε, μεταρρύθμιση της δημόσιας δίκησης που είναι θεμελιώδη. Και επίσης τονίζει ότι αυτά που ζητάμε από την Βοσνία Ζεγοβίνη είναι αυτά που ισχύουν για όλα τα άλλα υποψήφια κράτη-μέλη. Θέλουμε να στηρίξουμε τη χώρα στην πορεία της προς την ένταξη. Το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα για τη χώρα αυτή. Από την άποψη αυτή το βασικό θα είναι οι κυβερνήσεις σε κάθε επίπεδο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να σχηματιστούν. Για την Τουρκία που είναι εταίρο κλειδί για την Ελλάδα. Ο διάλογο και η συνεργασία σε ουσιώδει τομεί κοινού συμφέροντο συνεχίζεται. Αυτό συμπεριλαμβάνει ουσιώδη συνεργασία για τη μετανάστευση και τη στήριξη που δίνουμε για το θέμα των προσφύγων. Όμω η Τουρκία έχει συνεχίσει να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίσει να συνεχίζει να ε, έχει υπαναχωρήσει στο κράτος δικαίου και δεν υπάρχει στο πολιτικό σύστημα επαρκής ισορροπία και έλεγχη. Αυτό προεκλήθη και από τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Τον Ιούνιο του 2018 το Συμβούλιο ομόφωνα τόνισε ότι οι διαξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας έχουν βαλτώσει και δεν μπορούν να ε, κλείσουν ή να ανοίξουν περαιτέρω κεφάλαια. Η αξιολόγηση αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είναι το τελευταίο πακέτο διεύρυνσης που θα σας παρουσιάσω. Γι' αυτό επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους από εσά που είναι πολλοί που προσπάθησαν να προωθήσουν την ε, διεύρυνση της Ένωσης και εδώ και στο Στρασβούργο τα συζητήσαμε πολλές φορές πολλοί από εσά πήγατε επανειλημμένα στη χώρα τις προσεγγίσατε, συζητήσατε με τους λαούς και συμβάλατε σε πολλά από τα επιτεύγματα Πρέπει να τονίσω ότι πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι για όσα πετεύχθησαν. Φυσικά πολλά υπολείπονται ακόμη, αλλά αυτά που επιτύχαμε δεν θα ήσαν δυνατά παρά μόνο χάρη στη συνεργασία μας. Χάρη στην θαυμάσια συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και άλλων θεσμικών οργάνων. Αλλά πυρήνας ε, της πρόοδου ήταν η θαυμάσια συνεργασία μας και η ισχυρή σας δέσμευση. Γιατί δεν είναι μόνο μια στρατηγική επένδυση αυτό για το μέλλον της ε, περιοχής. Τονίζω και πάλι ότι είναι προς το συμφέρον και το δικό μας, της Ένωσης. Να έχουμε η περιοχή αυτή να είναι τμήμα της Ένωσης. Γιατί ανήκει στην Ένωση. Ήδη. Αλλά πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι χώρες αυτές. Ευχαριστώ για όλα όσα κάνατε και δεν ξέρω αν έχετε επανεκλεγεί, αλλά ιδιαίτερα σε όσους αποχωρούν από το Κοινοβούλιο, θέλω να πω ότι είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχίσετε να ενδιαφέρεστε και να, και να εργάζεστε για τα θέματα αυτά και ίσως θα βρούμε τρόπους για να συνεχίσουμε τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων γιατί όλοι πρέπει να βοηθήσουν, να στηρίξουν την προσπάθεια των χωρών αυτών στο κοινό μας ταξίδι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Johannes Hahn. Αγαπητέ Ζωχάνες Χάν, καταρχάς και νομίζω εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής μας, σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική σας δουλειά για την πολιτική της γειτονίας και της διεύρυνσης και για την εξαιρετική συνεργασία μας με την Επιτροπή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα 35 λεπτά χρόνο για να έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα για το ποιο έχει το λόγο και για πόσο χρόνο. συντονιστέ δύο λεπτά ο καθένα, αλλά εάν είναι ταυτόχρονα κάποιο και εισηγητή και ε, συντονιστή, μπορεί να έχει τρία λεπτά. Θα είμαι λοιπόν ε, ε, εξαιρετικά αυστηρό σήμερα. Και ο λόγο των Κρίστιαν Πρέντα, που είναι και τελευταία του συνεδρίαση στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και δεν είναι και μόνο συντονιστή, αλλά και εισηγητή. Τρία λεπτά. Ναι, να δούμε. Δέκα χρόνια χρειάστηκαν για να πάρω τρία λεπτά. Ε, καταρχάς, να πω ότι είναι πολύ θετικό ότι εγκρίθηκε το πακέτο της διεύθυνσης παρά το ιδιαίτερο πρόγραμμα εξαιτίας των ευρωεκλογών. Ελπίζω εν γέννη η πλειοψηφία υπέρ της Ευρώπης που θα δημιουργηθεί σε αυτό το κοινοβούλιο να συνεχίσει να προωθεί την ε, πορεία προς την Ευρώπη των Δυτικών Βαλκανίων όπως έχει γίνει ως τώρα, όπως κάναμε εμείς. Νομίζω η Επιτροπή μας τα δέκα τελευταία χρόνια διαρκώς ε, έδειχνε ότι είναι υπέρ αυτής της πορείας και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να στηρίξουμε την κάθε μια χώρα ξεχωριστά. Ιδίω τι φιλευρωπαϊκέ εκεί δυνάμει, ώστε να προχωρήσουν και σε δύσκολε στιγμέ. Νομίζω ότι αν δεν προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, θα ε, καταστεί δύσκολο να παραμείνουμε αξιόπιστοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, στο Συμβούλιο του Ιουνίου θα πρέπει επιτέλους να εγκριθεί η απόφαση να εναρθούν οι διαπραγματεύσεις με την ε, Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Νομίζω ότι είναι ανάγκη, επιτακτική. Του ζητήσαμε να κάνουν κάποια πράγματα πριν από ένα χρόνο, τα έπραξαν. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να επιβεβαιώσουμε την ποιότητα της εργασίας τους. Ως εισηγητής για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, εκφράζω την ε, ικανοποίησή μου για την ε, έκδοση της γνωμοδότησης για την ε, υποψηφιότητά τους για τη χώρα αυτή. Χώρα που, έγκριση μάλλον που συνοδεύεται από μια διεξοδική έκθεση αξιολόγησης. Πριν από πέντε χρόνια άρχισα να εργάζομαι για το θέμα της Βοσνίας. Δεν ήταν ακόμη υποψήφια χώρα. Την υποψηφιότητα δυσκολευτήκαμε να την προωθήσουμε για να βρεθεί κάποια λύση. Σήμερα λοιπόν επιτέλους έχουμε θετική τοποθέτηση από την πλευρά της Επιτροπής για την υποψηφιότητα αυτή. Ελπίζω και στο Συμβούλιο λοιπόν όλοι οι υπεύθυνοι να τα δουν αυτά με προσοχή και να καταλάβουν ότι είναι τεράστια ανάγκη για τη χώρα αυτή να της δοθεί αναγνώριση στο καθεστώς υποψηφιότητας. Και ως προς την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη ότι έχει πάρει τη σωστή πορεία προ την Ευρώπη και να υπάρξει σαφήνεια στο τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει. Γιατί όπω και η Ευρω... ο Επίτροπο μα είπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει κάποιε προτεραιότητε για τη δημοκρατία και τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να δούμε όλο το θέμα τη μεταρρύθμιση του διοικητικού μηχανισμού. Για τι αρχέ τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, λοιπόν, είναι η στιγμή να λάβουν το καθεστώ υποψήφια χώρα ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει και να ε, υπάρξει κάποια επιτάχυνση στο να απαντήσουν στα ανοιχτά ερωτήματα που παραμένουν. Ήθελα ολοκληρώνοντα, αγαπητέ Γιωχάνη Χάνα, να σε ευχαριστήσω για τι τεράστιε προσπάθειε που έκανε κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία και για όλο τον συντονισμό των προσπαθειών μα. Ευχαριστώ, Κρίστιαν Πρέντα. Τώρα στου σοσιαλιστέ και δημοκράτε, ε, η Κάτι Πύρη, εκ μέρου τη ομάδα. Είναι και η συγγήτρια για την Τουρκία. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία Πιτρόπεχάν, Πεχάν, αγαπητοί συνάδελφοι. Αντικαθιστώ σήμερα τον συντονιστή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τον κύριο Φλέκινστον, για την τελευταία συνεδρίαση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι Σοσιαλιστέ και οι Δημοκράτες υποστηρίζουν ακράδαντα τη διαδικασία διεύρυνση, ε, που είναι προ όφελο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των υποψηφίων χωρών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τι ε, δεσμεύσει τη, αλλά είναι αξιοκρατική η διαδικασία. Κάθε υποψήφια χώρα λοιπόν θα πρέπει να αξιολογείται βάσει των μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει. Και στη νέα θητεία η ομάδα μου θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φυσικά ο ρυθμό θα εξαρτάται από την κάθε υποψήφια χώρα. Είδαμε λοιπόν σοβαρέ επιτυχίε τα τελευταία πέντε χρόνια. Η συμφωνή των Προσπών που επέλυσε το θέμα τη ονομασία μεταξύ Ελλάδα και Βορρή Μακεδονία. Και αυτό αποδεικνύει εκ νέου ότι η διπλωματική οδός είναι η πλέον ενδεγμένη. Και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσουν κατά πόσον θα ξεκινήσουν διαδικασίες ε, για την διαβρύνση της με τη Βόρεια Μακεδονία και την ε, Αλβανία. Θα είμαστε υποθετικοί και για τις δύο χώρες, αλλά θα, προσπαθού, θα προτιμούσα να μην το είχε υποβάλει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πακέτο, γιατί είναι αντίθετο αυτό με την αρχή ότι θα πρέπει να υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια βάση χώρας. Αλλά παρ' όλα αυτά δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος για να καθυστερήσει η διαδικασία, μιας και τα κριτήρια πληρούνται και για τις δύο χώρες. Αυτό ελπίζω ότι θα παρατρύνει και τη Βοσνία Ριζεγοβίνη και το Κωσυφοπέδιο να ξεκινήσουν νέο γύρο σοβαρών μεταρρυθμίσεων προκειμένου στην μεραντική θητεία να δοθεί καθεστώς υποψηφίων χωρών σε όλες τις χώρες των Βετικών Βαλκανίων. Για το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τη δική τους ε, προθυμία να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις. Και συνολικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε σημασία στην μειούμενη ε, χώρο που έχουν τα ε, κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωση στι περιοχέ αυτέ. Και τέλο, στα Δυτικά Βαλκάνια έχει σημασία να συνεχιστεί και να διευκολύνεται η διαδικασία τη Πρίστινα σε ό,τι αφορά την εξομάλυση των σχέδιων μεταξύ σερβία και Κωσυφοπεδίου με κάλυψη όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Για την Τουρκία να πω δύο λόγια. Δεν έχω ακόμα διαβάσει την έκθεση, αλλά ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα έκθεση δεν θα έχει κάνει μία απλή καταγραφή των γεγονών Θα έχει διατυπώσει, ελπίζω, και μία στρατηγική για το πώ θα προχωρήσουμε, γιατί η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σαφή. Με την κυβέρνηση αυτή δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε διαπραγματεύσει για προσχώρηση αλλά παρόλα αυτά είμαστε αλληλέγγυοι και είμαστε στη διάθεση του λαού της Τουρκίας για τους δύσκολους καιρούς που περνάνε. Ακούμε διάφορες ε, κατηγορίες ε, για την κατάσταση που επικρατεί στην φυλακή, για την κατάσταση των Κούρδων που έχουν σταματήσει την απεργία πείνας. Και τέλος ε, είδαμε ότι ακόμα και ο τελευταίος πυλώνας στις δημοκρατίες της Τουρκίας, οι ελεύθερες άμεμπτες εκλογές, διακυβεύτηκαν με την διαδικασία για την εκλογή του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Απευθύνω λοιπόν έκκληση να αποσταλεί για τις 23 Ιουνίου μια έκτακτη αποστολή παρακολούθηση των εκλογών στην ε, Τουρκία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Χαν για την εξαιρετική συνεργασία τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια και καλή τύχη στο μέλλον. Σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι πήρε, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα να δώσω το λόγο στον Τσάρλ Στανοκ, ο οποίος είναι συντονιστής ε, και εισηγητής για το Μαυροβούνιο. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ και μια και θα αυτή η τελική μου, η τελευταία μου παρέμβαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε για το θέμα τη διεύρυνση. Ω εισηγητή για το Μαυροβούνιο τελευταία δέκα χρόνια, καλωσορίζω τα θετικά σα σχόλια, Επιτροπή Αχάν, για την πρόοδο που σημείωσε η χώρα. Ένα μόνο κεφάλαιο μένει να ανοίξει σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνιστικότητα και φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνει την προσοχή τη στο πώ θα κλείσουν τα κεφάλαια αυτά και προφανώς υπάρχει ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα του κράτους και του δικαίου στα κεφάλαια 23 και 24. Στην έκθεση, στο πακέτο μάλλον για τη διεύρυνση του 2018, συστήσατε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει με τις υποψήφιες χώρες Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Με την Συμφωνία των Πρεσπών, για την οποία πρέπει να πω ότι ήμουν περήφανος που συνυπέγραψα ε, τη συμφωνία με τον ε, Πρωθυπουργό Τσίπρα και φαίνεται ότι πλέον τίποτα δεν εμποδίζει την οδό και την πορεία της Βόρειας Μακεδονίας ε, και τις διαπραγματεύσεις με τη χώρα αυτή. Ελπίζω να υπάρξει κάποια κινητοποίηση μέχρι το τέλη του 2019. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτές, ε, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα σε ό,τι αφορά τη γενικότερη ατζέντα της διεύρυνσης. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι επιλογή. Θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί αναγκαιότητα, κάτι το αναπόφευκτο και όταν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει για τη διαμόρφωση τη νέα επιτροπή, ε, θα πρέπει να δοθεί μία έμφαση στον τομέα αυτό. Αν θέλουμε λοιπόν να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να υπάρχει αμετακίνητη στάση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για όλους τους πολίτες, για όλες τις χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν. Και τέλος, να δώσω το θέμα της χρηματοδότηση. Ε, χρηματοδότησης συνταξιακής χρηματοδότησης ε, και ιδιαίτερα του τρίτου σκέλους σε ό,τι αφορά και την επιτεύξη τελευταίας διαρρύθμισης ε, με το Συμβούλιο τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω λοιπόν να επαναληφθεί αυτή η ισχυρή δέσμευση για τη διαδικασία διεύρυνσης. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλους τους υπαλλήλου για την συνεργασία τους και την υποστήριξή τους στα 18 χρόνια της ε, θητείας μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Τσάρλ, για την συμβολή σου και για την καταπληκτική εργασία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στην Επιτροπή μα. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Έντουαρτ Κούκαν. Δύο λεπτά. Είναι πρόεδρος της ε, ομάδα εργασία για τα Δυτικά Βαλκάνια και πρόεδρο τη αντιπροσωπη σχέση με τη Σερβία και νομίζω ότι είναι και η δική σα τελευταία συνεδρία. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ για όλα όσα κάνατε τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίτροπε Χάν, νομίζω ότι ορισμένες φορές ε, τα παροχημένα κλισέ μπορεί να φαίνονται σαν ειλικρινείς δηλώσει. Και θέλω να πω λοιπόν ότι ήταν για μένα τιμή και ευχαρίστηση η συνεργασία μαζί σας. Η έκθεση που παρουσιάζεται σήμερα, Επίτροπε, αναμενόταν από πολλούς με πολύ ενδιαφέρον. Ήταν το θρίλερ της χρονιάς. Η πρώτη μου αντίδραση σε αυτά που άκουσα είναι θετική. Θέλουμε οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων να κάνουν άλλο ένα βήμα προς την ένταξη. Γι' αυτό θεωρώ ότι και η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν αυτά τα επόμενα βήματα όπως προτείνεται. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα θετικά Υπήρξε πρόοδρος ε, προς την ένταξη, αλλά παράλληλα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα. Καλύτερη πρόοδος. Νομίζω ότι χρειάζονται τη συνεχή βοήθειά μας και προσοχή. Έχει κάνει πολλά η Βόρεια Μακεδονία, αλλά πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να γίνουν πραγματικότητα οι βάσεις που έχουν θέσει. Με την Αλβανία είναι, υπάρχει μεγάλη ένταση στο εσωτερικό. Έχουν τοπικές εκλογές ε, στις 30 Ιουνίου και να πόκειται ε, στην πολιτική ηγεσία της χώρας να ξεπεράσει τα μικροκομματικά συμφέροντα και να λάβει τις αποφάσεις που θα εξυπηρετήσουν το λαό της Αλβανίας, που πραγματικά του αξίζει το καλύτερο. Σωστά είπατε ο, τι αναμέναμε από τους εταίρους μας. Σωστά τα απαριθμίσατε. Αλλά και εμείς ε, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πιο θεαματικό, να ξαναδούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα, για να ασκήσουμε θετική πίεση στις χώρες αυτές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί αν δεν το κάνουμε, ανησυχώ και φοβάμαι ότι θα διαβρωθεί η αξιοπιστία μας, το κύρος μας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα θέματα ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έντουαρτ Κούκαν. Οι υπόλοιποι μόνιμοι συγκητές 1,5 λεπτό καθένας. Πρώτος, ο Ιβο Για τη Βόρεια Μακεδονία. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η περιφερειακή σταθερότητα μιας πολύ σημαντικής ε, και πολύ ευαίσθητης περιοχής. Αν θέλουμε σταθερότητα στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε σταθερότητα και εδρεωμένη δημοκρατία στα Δυτικά Βαλκάνια, συνολικά. Στηρίζω την έκθεση. Και σας ευχαριστώ, Επίτροπε Χάν, για την εργασία σας. Θαυμάσια δουλειά. Και προσωπικά δώσατε πολλά για να βοηθήσετε να επιληθούν πολλά προβλήματα. Ως εισηγητής για την Βόρεια Μακεδονία τονίζω ότι το θέμα δεν είναι τι έχει επιτύχει η ίδια η χώρα. Είναι και τι υποσχέσεις της δώσαμε. Τι δεσμεύσεις αναλάβαμε. Δεσμευθήκαμε, υποσχεθήκαμε στο λαό και στους πολιτικούς της Βόρειας Μακεδονίας ότι εάν, εάν ε, σέβονται τα υπεσχημένα, εάν είχαν νέα προσέγγιση στις σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες, εάν ε, επετύχαναν ένα καλό συμβασμό με την Ελλάδα, θα έπρεπε να ανταμυφθούν. Οι δεσμεύσει θα έπρεπε να γίνουν σεβαστές. Και τελειω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει κάθε αξιοπιστία στην περιοχή, όχι μόνο στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά συνολικά στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ιβο Βάγκλ. Ο Ιγκοσόλτες δεν είναι εδώ, οπότε να δώσω το λόγο στον Ντέιβιντ ε, Μακάλιστερ, που είναι ο μόνιμος συζητητής για τη Σερβία. Ο συζητητής λοιπόν για τη Σερβία διαπίστωσα ότι η χώρα έχει επιτύχει αποτελέσματα, ιδιαίτερα για την μακροοικονομική σταθεροποίηση και αυτό ωφέλησε φυσικά και το λαό. Αλλά παράλληλα, πιστικές μεταρρυθμίσεις χρειάζονται ακόμη στη Σερβία, ιδιαίτερα στο δικαστικό τομέα, την καταπολέμηση διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων και μια άλλη τρομερή πρόκληση είναι ο διάλογος για την εξομάλυση των σχέσεων με το κοσφοπέδιο πρέπει ταχαίως να επανέλθουν στο διάλογο και να καταλήξουν σε νομικά δεσμευτική συμφωνία. Προχωράει λοιπόν η Σερβία προς την ένταξη. Ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων όμως εξαρτάται από το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στην Σερβία σε τομείς κλειδιά. Πολλά υπόθηκαν από συναδέλφους από διάφορες πολιτικές ομάδες. Να προσθέσω και κάτι. Όχι όπως προηγούμενα χρόνια, Είμαι πεπισμένος ότι αυτή τη φορά οι εκθέσεις δεν διέρευσαν προς τα μέσα. Οπότε είμαστε οι πρώτοι που ακούσαμε. Αυτό είναι θαυμάσιο. Ακούσαμε τι έχει γίνει. Και αυτό είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο. Ας ε, ελπίσουμε ότι θα γίνει παράδοση για τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα πέντε χρόνια. Και ενημερώθηκα ότι λάβαμε μέσω email το, τις εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ενάμιση λεπτό πιστεύω. Και τώρα, και τώρα ο Ιωάννη Χάν πρέπει να πάει σε μια διάσκεψη τύπου. Οπότε πρέπει να φύγει στι 12.35. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη. Λοιπόν, ποιοι έχουν στήσει το λόγο. Μισόβκο, Ντέλη, Γιακοντζάρη, Γκόμε, Οστρεβίτσιου, Χατζηγεωργίου και Μπίλτ. Μπορκέτσιο επίση και, και Σελίμοβιτ. Ωραία, κλείνει ο κατάλογο. Ένα λεπτό ο καθένας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε για τη θετική σας τοποθέτηση για την έκθεση της Βοσνίας Αρζεγοβίνης. Για την Κροατία είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μας ενδιαφέρει η ειρήνη και η σταθερότητα και σε σχέση με τα ε, σύνορά μας ε, προς τη Βοσνία Ριζεγοβίνη και γενικότερα σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ' αυτή την έννοια και βάσει της παρατηρήσεις και του Προέδρου μας πρέπει να πω ότι ε, δεν μπόρεσα να διαβάσω την έκθεση αλλά πραγματικά θα εκτιμούσα το να δοθεί προσοχή στην, ε, στο σεβασμό των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου και αυτό να τεθεί ω προπόθεση στο ίδιο επίπεδο με την αιρεσιμότητα για το σεβασμό των ε, αποφάσεων του Δικαστηρίου στο Στρασβούργο διότι η σχετική αστάθεια στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει να κάνει και με την κακή λειτουργία του εκλογικού νόμου. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξει για να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα και εντό τη χώρα τη ίδια. Ε, και να προσθέσω ότι το θέμα της ε, επιρροής που ασκείται σε άλλες, από άλλες χώρες, ε, ιδίως από την Κίνα, στην περιοχή, μέσα σε αυτή τη χώρα, είναι ένα θέμα. Πρέπει να το λάβουμε προσεκτικά υπόψη. Κατά την κατάρτιση των αποφάσεών μας για την Βοζία Ρεγοβίνη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Σόφκου, κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ. Ανοιχτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ωραίο να ολοκληρώνουμε αυτή τη θητεία με τη συζήτηση της ιστορικής απόφασης. Η ευρωπαϊκή πολιτική της διεύρυνσης ως τώρα έχει υπάρξει μια από τις πλέον ε, επιτυχημένες ε, ε, δράσεις της εξωτερικής μας πολιτικής. παρόλο που έχει προκαλέσει και τόσα αρνητικά συναισθήματα, είτε από την κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μεμονωμένα σε επίπεδο κάποιων κρατών μελών. Πρέπει όμως να είμαστε συνολικά πολύ ε, ικανοποιημένοι με το επιτευγμά μας. Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ταυτόχρονα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό που λείπει είναι η συστηματική παρακολούθηση του πώ υλοποιείται αυτή η στρατηγική. Πέρσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ενέκρινε τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων και με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία. Αυτό έχει κάπως αποδυναμώσει και πλήξει την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, διεύρυνσης. Συνολικά όμως είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ συνάδελφε. Τώρα ο κύριος Πέτρα Αουστρεβίτσιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και Επίτροπε για την συνεργασία σας με την Επιτροπή μας. Σας εύχομαι κάθε καλή τύχη και ε, ανυπομονώ να ξανασυναντηθούμε στι αρχέ του φθινοπόρου. Ε, Προσυπογράφω στι δηλώσει σα ότι η πολιτική διεύρυνση είναι πολιτική σταθερότητα για τι συγκεκριμένε γεωγραφικέ περιοχέ και όλη την Ευρώπη. Οι χώρε διεύρυνση θα παραμένουν προτεραιότητα και την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ελπίζω ότι θα έχουμε ακριβώ το ίδιο επίπεδο συνεργασία και καλή συνεννόηση. Συνάδελφοι, σα ευχαριστώ ε, για τι συνεισφορέ σα στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ιδίω για τι χώρε σύνδεση και αυτέ που βρίσκονται στην ταξιακή πορεία. Η προοπτική θα πρέπει να παραμένει ένα ισχυρό κίνητρο για να εκτελούνται μεταρρυθμίσει εντός των χωρών. Ξέρουμε ότι όταν τους ζητάτε γίνονται αυτές. Θα πρέπει όμω να καταστεί σαφέ και από τη δική μου την πλευρά ότι η πολιτική διεύρυνση εμπνέει τις χώρε ε, βάσει των συμφωνιών ε, ένταξη να προχωρήσουν σε επιτυχημένη υλοποίηση πολιτικών στο εσωτερικό της χώρας. Επίτροπε υπάρχουν νέα μέσα που θα μπορούσαν να συνδράμουν τις χώρες να, να πράξουν αυτές τις μεταρρυθμίσει με τρόπο ομαλότερο. Ευχαριστώ κύριο Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Χάν. Ευχαριστώ και τον κύριο Χάν πάρα πολύ για όσα έχει κάνει ως τώρα, πάντα θετικός και πάντα ανοιχτός σε κάθε συζήτηση και ήθελα να το πω αυτό. Ε, υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν νομίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση εξωτερικής πολιτικής και αφορούν το ένα το Κόσοβο και τον άλλο το Κυπριακό. Είναι δύο μεγάλα προβλήματα άλυτα. Ε, ερχόμενος στο θέμα Τουρκία ασφαλώς, να υπομνήσω και εγώ αυτά που ήδη ελέγχθησα για πληροφορίες για βασανισμούς στις τουρκικές φυλακές, ακύρωση εκλογών αλλά νομίζω ότι υπάρχει και μια παραβίαση της συμφωνίας για το προσφυγικό, υπογραμμίζοντας ότι χιλιάδες μετανάστες έρχονται από την Τουρκία προς την Κύπρο. Και αυτό είναι καταγραμμένο και σε εκθέσεις της Κομισιόν. Και δεν μπορεί πλέον να είναι τυχαίο, είναι σκόπιμο. Το δεύτερο που έχω να πω, υπάρχει η επιδρομή της Τουρκίας στην περιοχή Τη αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, επικαλούμενη μάλιστα την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, την ώρα που είναι η μόνη χώρα που δεν υπογράφει αυτή τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας στα Ηνωμένα Έθνη. Και ακούγεται περίπου ως επιχείρημα λίγο αστείο. Κλείνω γιατί έχω ξεπεράσει τον, τον χρόνο, αλλά ήθελα μια απάντηση σε αυτά Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Επίτροπε. Τα μέλη τη αντιπροσωπείας τη Βοσνία Ερζεγοβίνης. Το θέμα λοιπόν είναι να ρωτήσω τα... για το θέμα το οποίο αναφερθήκατε στην ανακοίνωση τύπου σε ό,τι αφορά τις χώρες αυτές και την διαδικασία της κίνα του δρόμου του μεταξιού. Οι επενδύσεις, ε, οι κινέζικες, έχουν ε, υπονομεύσει την επικυριαρχία των χωρών. Και το θέμα της ε, οικονομικής ε, βιωσιμότητας είναι επίσης σημαντικό. Μιλάμε για 900 δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά την δημιουργία αυτοκινητοδρόμου. Και από την άλλη, η συνοχή με τους ευρωπαϊκούς στόχους των επενδύσεων αυτών για θέματα περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η Βοσνία Ερζεγοβίνη τον περασμένο Απρίλιο έκανε μια σύμβαση με κινησική εταιρεία για την ανακαίνιση με εργοστασίου άνθρακα. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν των Βαλκανίων με την Κίνα πιστεύετε ότι συνάδει με τις ε, ευρωπαϊκές βλέψεις της περιοχής και τι θα συνέπειες θα έχει στην διαδικασία διεύρυνσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπίλτ. το τέλει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Επίτροπο Χάν για την δουλειά που έχει κάνει και τη μεγάλη δέσμευσή του. Δεν αναφερθήκατε όμως στα κεφάλαια και στα κεφάλαια που θα ανοίξουν. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για την Σερβία και το Μαυροβούνιο, τι κεφάλαια και ποια κεφάλαια θα μπορούσαν ενδεχομένω να ανοίξουν. Κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι υπάρχει οποιοδήποτε πλουτική να λυθεί το θέμα μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου. Γιατί προφανώς ε, οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της κρίσης που επικρατούν και η μόχλαυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποφέρουν καρπούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει κάποιον άσο κρυμμένο, κάποιο τζόκερ. ή θα αναλάβουν τα ενία τα κρατημέλη όπως έχει κάνει η Γαλλία και η Γερμανία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ντέλη. Η κυρία Γκόμες. Ναι. 15 μέλη 15 χρόνια είμαι μέλο τη επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και δύο υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ασφάλεια, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά πάνε χέρι-χέρι. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω, Επίτροπε, γιατί αυτή η σταθερότητα δεν αποτελεί αυτό σκοπό και αυτό αξία. Όχι βέβαια, αν έχει ω σκοπό την διαιώνιση της καταπίεση. Οι αξίε μα ποιε είναι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κρατοδικαίο. Και γι' αυτό ακριβώς με τα Δυτικά Βαλκάνια και με την Τουρκία το βασικό ζητούμενο για μας, η βασική στρατηγική επένδυση θα πρέπει να είναι στην κοινωνία των πολιτών. Το ρόλο που μπορεί να τετραματίσει η κοινωνία των πολιτών σε ό,τι αφορά και τις κυβερνήσεις που έχουν την εξουσία, προκειμένου για να βελτιωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε τι γίνεται στην ε, Τουρκία οι δικαστές και κυρίως οι γυναίκες οι δικαστές έχουν φυλακιστεί υπό φρικτές συνθήκες. Εγώ ως πρώην διπλωμάτης πρέπει να βγω να μιλήσω για τους διπλωμάτες. Χτες είχαμε μια φρικτή αποκάλυψη για διπλωμάτες που έχουν μπει στις φυλακές της Τουρκίας. Δεν μπορεί να σιωπήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτόν. Ευχαριστούμε την Άννα Γκόμες, λέει ο πρόεδρος Σελίμοβιτς. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο και με πάσα ειλικρίνεια κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά σε πολύ δύσκολους καιρούς. Και αυτούς τους καιρούς λοιπόν που διανύουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς λοιπόν για το θέμα αυτό και να πω και στους συναδέλφους να... ότι οι κυρία έχουν αλλάξει. Τα κόμματα τα φιλελεύθερα τα οποία ήταν υπέρ της διευρυνσής που την έβαλαν στην ατζέντα ε, εδώ είναι τα κόμματα τα οποία κέρδισαν με μεγαλύτερη διαφορά εδώ στις εκλογές. Αυτό λοιπόν θα πρέπει κάπως να μεταφραστεί, να αποτυπωθεί στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επόμενη θητεία. Προσπαθήσαμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτή την ατζέντα ακόμα και με κόμματα και με πολιτικές ομάδες προστατευτικές. Προσπαθήσαμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτή την ιδέα της Ευρώπης που προστατεύει, αλλά τώρα πλέον αυτοί που ουσιαστικά νίκησαν είναι οι φιλελεύθεροι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτυπωθεί στην ατζέντα της διεύρυνσης. Όχι μόνο γιατί υπάρχει θέμα ασφάλειας, υπάρχει θέμα ειρήνης στην ε, περιοχή, αλλά επειδή αυτό επιθυμούν οι εκλογείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τελευταίο ο κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τις 24 Μαΐου έχω θέσει ένα επίμονο ερώτημα και Επιμένω γιατί είναι ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει σύγχυση και αστάθεια σε κάποιες από αυτέ τι χώρες. Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κόσοβο, Αλβανία. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα θέματα της μετανάστευση και ε, ακόμα και με την εμπορία ανθρώπων για τη δουλειά που κάνουμε εμεί και την απάντηση που θα μου δώσετε. Θα πρέπει ε, να προασπιστούμε τους εαυτού μα από αυτά τα προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν μια τοποθέτηση σαφή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να λάβω το θάρρο να να επισημάνω ότι τέτοιε απορίες είχαμε θέσει και στο παρελθόν και από την ΕΝΕΦ είχαμε υπογραμμίσει και του κινδύνου και το ρίσκο που προέκυπτε από την συμφωνία με την Τουρκία και την προοπτική τη συνεργασία μας μαζί της. Τα αποτελέσματα δεν ήταν και λαμπρά. Δεν θέλω λοιπόν να ακουστώ ω προφήτη, αλλά πραγματικά ε, αυτά έρχονται να κολλήσουν με τι ανησυχίε που είχα ε, εκφράσει. Και ο Νοστράδαμος ε, το είχε πει δεν ξέρω αν δεν θα βρεθούμε προ μεγάλων εκπλήξεων όταν προσχωρήσουν αυτές οι χώρες, αυτοί οι λαοί και αν θα έχουμε και την όθηση που θέλουμε και είδαμε να προκαλεί τόσα προβλήματα σε χώρες όπως η Ιταλία. Καλό κουράγιο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, Επίτροπε Χάν. Έχετε χρόνο για να απαντήσετε και να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε θα υπάρξουν κι άλλε ειδικότερε σε ένα χώρα και με μεγάλη χαρά να ξανασυζητήσουμε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σας ευχαριστήσω όλους για τα θετικά σα σχόλια και την έκφραση της ικανοποίησής σας για τη δουλειά μας. Θα πω όμως και θα επαναλάβω και θα ξαναπώ ότι όλα μας τα επιτεύγματα δεν θα είχαν ε, καταστήνατα χωρίς τη δική σας αφοσίωση τη σκληρή σας δουλειά και την ε, άοκνη εργασία σας. Πρέπει να το τονίσω. Νομίζω ότι αφήνουμε μια πολύ θετική κληρονομιά για την επόμενη θητεία και του επόμενου που θα αναλάβουν στην Επιτροπή αυτή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Φυσικά θα υπάρξουν κάποια σημεία όπου η επόμενη γενιά, για να το πω έτσι, θα πρέπει να τα επεξεργαστεί καλύτερα. Για κάποια από τα σχόλιά σας τώρα, από τις παρεμβάσεις σας. για τα νέα μέσα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε λόγο για νέα μέσα. Αλλά όπω ήδη είχαμε συζητήσει για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, η ιδέα να γίνει αλλαγή στην δομή της πολιτικής ώστε να μην έχουμε χαρτοφυλάκιο αναχώρα πλέον, αλλά χαρτοφυλάκιο αναθέμα ώστε να μην προκύπτει ανταγωνισμός, μάλλον να προκύψει κάποιο είδους άμυλα μεταξύ των διαφορετικών χωρών για να αντιμετωπίσουν παρόμοιες προτεραιότητες σε μια κοινή διαδικασία. Βεβαίως, στην ε, τελική φάση θα πρέπει όλοι να οκληρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις. Αλλά θα μπορούμε να θέτουμε σε συγκεκριμένε χώρες προτεραιότητες και να υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία έτσι, ώστε να προκύψουν και περισσότερες δυνατότητε για τέτοια ευγενή άμυλα. Και ε, ένα θετικό ανταγωνισμό. Ήταν ένα πολύ θετικό εργαλείο για να παροτρύνουμε την ε, εντατικότερη δουλειά στην όλη περιοχή. Δεύτερον, νομίζω ότι αν σωστά καταλάβατε κυρία Γκόμες, πράγματι η σταθερότητα δεν θα πρέπει να παρερμηνεύεται ως ε, απλώς σταθεροποίηση, παγίωση κάποιου καθεστώτος. Είναι μία βάση ένα εφαλτήριο από το οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάπτυξη. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν αρμονικές ε, σχέσεις και συνεργασία του οικονομικού τομέα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και όλα τα υπόλοιπα. Διότι το χειρότερο που μπορούμε να δούμε να συμβαίνει είναι να διαφεύγουν κάποιοι από τις διάφορες χώρες και πρέπει να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες. Δεν είναι προς όφελός μας κάτι τέτοιο. Θα πρέπει στους νέους να δώσουμε ελπίδα να ξέρουν ότι μπορούν να λάβουν την απαραίτητη μόρφωση και να έχουν προοπτικές και μέλλον στην ίδια τους τη χώρα. Αν αυτό συμβαίνει, είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα έχει ε, επίδραση στο σύνολο της αναπτύξής μας. Για την κοινωνία των πολιτών λοιπόν πρέπει να λάβουμε μέτρα και για το μέλλον. Αλλά έχουμε πολλά θετικά κίνητρα για να συμμετάσχουν περισσότερο στη διαμόρφωση της πολιτικής και την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και να μην μείνουν στο περιθώριο, ζητώντας από εμά τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να παρέμβουμε για να τους σώσουμε για κάτι. Αυτό είναι κάτι που έθεσε και η κυρία Μπίλντερ. Στην περίπτωση του δανείου για το εργοστάσιο που λειτουργεί με λιγνίτη. Δεν μας αρέσει η ιδέα αυτή. Συζήτησα ωστόσο με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών του περιβαλλοντικού χώρου και θα πρέπει να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες τους. Ήδη την περασμένη εβδομάδα το συζήτησα και μίλησα με κάποιους που ως εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, περιβαλλοντικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ήρθαν ε, για τη συνεδρίαση αυτή από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι καν από τις χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν καθαρή ενέργεια ας πούμε, παρά άλλες συμβατικότερες μορφές. Πρέπει να γίνει λοιπόν πολλή δουλειά να δούμε ποια είναι τα παλιά γενιά και τα νέα γενιά κριτήρια για την, για την προσχώρηση και ούτω καθεξή. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγέ. αλλά πρέπει να υπάρξουν και τα μέτρα, ώστε ο κόσμο στι διάφορε χώρε να μπορεί να έχει κάποιο λόγο στο εάν δημιουργηθεί κάποιο εργοστάσιο για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, να προσφέρει και περισσότερε δυνατότητε για την εργασία και την απασχόληση σε μια τέτοια περιοχή, για τι επενδύσει από την Κίνα και άλλε χώρε. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον σεβασμό του δικαίου ανταγωνισμού των δημοσίων προμηθειών, για τη διαφάνεια, την βιωσιμότητα των επενδύσεων και το τι σημασία μπορεί να έχει αυτό για τις ε, επιμέρους χώρες και τους ανθρώπους της οικογένειας εκεί, τα νοικοκυριά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της ευρωπαϊκής στήριξης και της στήριξης από αλλού. Μας νοιάζει, μας νοιάζει τι συνέπειες θα υπάρξουν από τη στήριξή μας. Γι' αυτό δεν βιαζόμαστε να δώσουμε ε, κάποιο, δάνειο λόγου χάρη. Το παρέχουμε ως ποσό, αλλά κοιτάζουμε να συνοδεύεται και από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να είναι ξεκάθαρο ε, τι απαιτήσει έχουμε από την πλευρά του οικονομικού τομέα και της κοινωνίας και να γίνονται σεβαστά και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ή να υπάρχουν ίσοι κανόνες ανταγωνισμού για την συνεργασία που παρέχουμε και στις υπόλοιπε ε, ευρωπαϊκές χώρες. Είναι κάτι που θα μας υποσχολήσει εντονότερα στο εγγύς μέλλον. Για το θέμα του διαλόγου. Ένα περαιτέρω παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να πάρει το πρόσωπο του πράσινου φως η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία για την άνοιξη των διαπραγματεύσεων. Είναι το ισχυρότερο κίνητρο, το καλύτερο επιχείρημα για τους υπολείπους ώστε να ξεκινήσει ένα τέτοιο διάλογο. Δεν είναι εύκολο ούτε για τη μια πλευρά ούτε για την άλλη. Χρειάζεται να υπάρξει θάρρος, τόλμη για να ξεκινήσει κανείς αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί στο τέλος της διαδικασίας θα χρειαστεί οπωσδήποτε ένας συμβιβασμός, κάποια συμβιβαστική λύση τη συμβαστική λύση, σίγουρα δεν θα την υποστηρίξουν 100% όλοι οι άνθρωποι στην Σερβία ή όλοι οι άνθρωποι στο Κωσυφοπαίδιο. Θα πρέπει όμω οι ηγετικέ μορφέ να ξέρουν ότι θα υπάρξουν θετικέ συνέπειε. Και οι συνέπειε θα πρέπει να είναι, οι επιπτώσει, ότι θα υπάρξει μια πορεία που θα ε, ανταμείψει την ε, διαδικασία προσχώρησης και τις προσπάθειες για την ευρωπαϊκή προσχώρηση. Γι' αυτό λοιπόν η ένωση διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία θα λειτουργήσει ως κίνητρο και για, τις, για τους ηθήνοντες που ασχολούνται με άλλα περίπλοκα ζητήματα και άλλες δυσκερείς καταστάσεις στην περιοχή αυτή. Είναι σημαντικό λοιπόν και να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τους υπολείπους. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί ένα θετικό σήμα προς τη μια ή την άλλη χώρα, ώστε να ε, παραδειγματιστούν και οι γύρω χώρες. Επίσης, για τα περαιτέρω ζητήματα και τις λεπτομέρειες. Θα έχουμε και άλλες συναντήσεις και συζητήσεις ε, αναχώρα. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω πολύ όλους τους ε, συναδέλφους που θα φύγουν από το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνετε από τον τέλειο Οκτωβρίου και μετά, αλλά εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω προσωπικώ ότι ό,τι και να κάνω θα παραμείνω αφοσιωμένο στο σκοπό αυτό, στην περαιτέρω ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων και στο μέλλον. Όταν έχει κάνει επενδύσει τόσο χρόνο και ενέργεια για ένα τέτοιο θέμα, δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να εργάζεται προς τον ίδιο σκοπό για να υπάρξουν και άλλες ε, θετικές ε, ε, και άλλα θετικά βήματα και επιτυχία και στο μέλλον. Ευχαριστώ και αντίο σας. Thank you. Ευχαριστούμε διάφορα. Η πρώτη μάλλον συνεδρίαση για σύνταξη σε σώμα θα είναι στις 8 Ιουλίου, μάλλον όχι στις 8 Ιουλίου, στις 10 Ιουλίου από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει όμως ακόμα επιβεβαιωθεί τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και πέρα στη συνεδρία σας.